για τα θέματα αυτά μέσα στο νομικό πλαίσιο που μας παρέχουν οι συνθήκες. Ευχαριστούμε. περούτη η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη στις 12. Προχωρούμε τώρα στην εξέταση της έκθεσης ΕΛΕΔΑ πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και ανάπτυξη πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναλάβει σε, ευρω... σε διεθνές επίπεδο να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο ε, για την ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων. Στο πλαίσιο ε, ε, της Συμφωνίας του Ελσίνκη έχει αναφερθεί πολλές φορές αυτό και πολλές φορές υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Πολύ συγκεκριμένα στις μη στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Eurolex και τη UPOL Μόνο το, ε, ε, ε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν, θέσεων που δεν καλύπτονται, που θα έπρεπε να καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι οι στόχοι μας ακόμη απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και γι' αυτό υπάρχει η έκθεση, κοινοβουλίας, του η έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη πολιτικοστατιωτικών ικανοτήτων. Το Κοινοβούλιο στην έκθεση αυτή διατυπώνει τη θέση του ότι οι πολιτικοστρατιωτικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ε, εξωτερική πολιτική μας και την πολιτική ε, ασφάλειας και άμυνας Καταρχήν ξεκινήσαμε από τους εμπειρικούς λόγους για τη δημιουργία μιας έκθεσης και είδαμε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία για την εξωτερική δράση και βάσει αυτών των στοιχείων διατυπώσαμε μια συγκεκριμένη έκθεση. Σε στρατηγικό επίπεδο καταρχήν θέλουμε να υπάρχει ε, μια ε, δομή μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων που θα είναι εξοπλισμένο με προσωπικό από τα κράτη-μέλη. Ε, συζητήσαμε ακόμη θέματα κινήτρων που θα προσφέρονται σε εθνικούς εμπειρογνώμονες για να συμμετέχουν σε τέτοιες ε, δραστηριότητες. Έχουμε συζητήσει επίση θέματα κατάρτιση και δημιουργία προσωπικού που θα ασχολείται με τα θέματα αυτά στο μέλλον. Ασχοληθήκαμε και με πολύ συγκεκριμένα θέματα για το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Υπάρχουν θέματα χρηματοδότηση αποστολών δημιουργία ενός ταμείου ε, ε, αρχικής προώθησης ε, και υπάρχουν και θέματα για τη διαχείριση κρίσεων και μελλοντική στενότερη συνεργασία αστυνομικών και αστυνομικών δυνάμεων. και υπάρχει γενικά ε, μέσα στην έκθεση το θέμα του πώ μπορούν να συνδυάζονται οι πολιτικές και στρατιωτικές δράσει, ώστε να μην υπάρχει διαχωρισμός καθαρά στρατιωτικών και καθαρά ε, πολιτικών ε, δραστηριοτήτων για το μέλλον των battle groups, των ε, μάχημων ε, μονάδων. Ε, έχουμε προτείνει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, έχουμε προτείνει στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών του όσων να αναπτυχθούν αυτά τα battle groups και να ενδυναμώσουμε τις ικανότητες αυτών των battle groups να αναλαμβάνουν πολιτικές αποστολές και να διαβρύνουμε το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των battle groups. Επίσης, στο πλαίσιο των, του προγράμματος πλαισίου ε, για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δυνατότητες που προσφέρονται και ε, για τις ε, τον εξοπλισμό διτής χρήσης για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρήση των δομών που ήδη υπάρχουν και για να έχουμε ε, δυνατότητες και στον τομέα των εναέριων μεταφορών και την καλύτερη συνεργασία σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων. Κυρίε και κύριοι, πιστεύω ότι με την πρωτοβουλία αυτή το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται τις ευθύνες που έχει σε αυτό το τομέα. Η έκθεση αυτή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έτυχε την ευρεία πλειοψηφία από όλε τι πολιτικέ ομάδε και νομίζω ότι δείχνει την μελλοντική κατεύθυνση για την πολιτικοστατιωτική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Διαδικασία Κατσιάη. Μόνο ένα. Ο κύριος Ζέγγεντ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι η πραγματική πολιτική και στρατιωτική συνεργασία. Εμείς θεωρούμε ότι όντως η πολιτικοστρατιωτική συνεργασία απαιτεί και τις δύο διαστάσεις. Η Ουγγαρία είναι καλό παράδειγμα διότι η Γκάρντα εμφανίστηκε ε, το 2007 και είδαμε πως ε, μπορούσε πως μπόρεσε να παρέμβει γρήγορα και σε σημαντικές αστικές μη στρατιωτικές δηλαδή πολιτικές δραστηριότητες υπήρξε ωστόσο αναγνώριση καμία αντί να αναγνωρίσει το πνεύμα θυσίας της ε, εθνοφρουράς, την διέλυσε η κυβέρνηση. Παρόμοιοι αντιοργανισμοί με το γκάλι υπάρχουν και αλλού. Αυτοί που θέλουν να μετάσχουν σε τέτοιες δράσεις ε, και θέλουν να βοηθήσουν ε, την συνεργασία θα πρέπει να προωθήσουν την συμμετοχή των ανθρώπων αυτών σε αντίστοιχε δραστηριότητε στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριο Εβενχάουζερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. οι πολιτικο στρατιωτικε ικανότητες ε, ήδη έχουν αναπτυχθεί, ιδιω. αν δούμε το κέντρο ανάλυσης ε, καταστάσεων, παραδείγματος χάρη. Εδώ έχουμε ε, σαφώς συνδυασμό πολιτικής και στρατιωτικής ικανότητας η ευρωπαϊκή δράση θα πρέπει στο εξωτερικό να εμφανίζεται μέσω και της πολιτικής της δράσης και έτσι να την χάνει αναγνώρισης. Ήθελα να πω κάτι το οποίο ήδη αναφέρθηκε και κάτι το οποίο ε, ε, με ενδιαφέρει και εμένα για την Ουγγαρία και το κόμμα Γιόμπιτς ε, που στην περιοχή των συνόρων με όπλα αναλαμβάνει την επιβολή της και νομίζω ότι αυτό είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι υπέρ της ευρωπαϊκής σκέψης. Ευχαριστώ. Eh, eh, eh, ο κύριος Ερενχάουζερ δέχεται να του τεθεί μια ερώτηση με μπλε Κοιτάξτε, να απαντήσω θέλω πρόεδρε σε αυτά που είπε ο κύριος συνάδελφος. Ψεύδι. Το Γιόμπικ δεν ούτε το Γιόμπικ ούτε η Γκάρντ έκανε τέτοιες πράξεις όπως αυτές που κατήγγειλε ο κύριος συνάδελφος, ούτε παραβίασε από τον νόμο. Αυτά είναι προπαγάνδα νεοφιλελεύθερη που θέλουν να, να πούν ότι το Γιόμπικ και η Γκάραντι είναι οι κακοί, που δεν έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο, είναι πάντα, ε, σέβονται πάντα τον νόμο. Ε, συγγνώμη, αλλά δεν είπα ότι ήταν ποινικού περιεχομένου η δράση τους. Είπα όμως ότι με καραμπίνες και με όπλα ε, βάδιζαν σε πορεία και νομίζω ότι από αυτού δεν μπορεί να φέρεται αντίρρηση. Ε, Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το λόγο τώρα έχει η Επίτροπος. Κύριε Δαμανάκη, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ στην έκθεση, δεδομένου ότι αυτό, αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση, εξαιρετικά σημαντική και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έλλαρ για την συνεισφορά του. Είναι χρήσιμη η έκθεση γιατί πολύ σωστά επικεντρώνεται στα βασικά στοιχεία της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας που αποτελούν και προτεραιότητα της Επιτροπής. Ασχολείται με τα βασικά στοιχεία που αφορούν την ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης κρίσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Η δημιουργία ε, της Ευρωπαϊκής ε, ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης αποτελεί ακριβώς αυτή την ε, ε αντίληψη. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος δημιουργεί αυτή την ε, υπηρεσία και οι σκοποί της ακριβώς κινούνται προς την κατεύθυνση της έκθεσης κυρίως με το να συμπεριληφθούν οι δομές της κοινή ασφάλειας, ε, και της ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας ε, στην ε, υπηρεσία αυτή. Στηρίζουμε απόλυτα την ανάπτυξη πολιτικών δυνατοτήτων ώστε να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ των πόρων. Οι, οι κατάλληλοι τρόποι είναι τώρα θέμα συζήτησης και μπορεί να προσκληθεί οι ειδικοί προς το σκοπό αυτό. Μέχρι τώρα αυτό δεν ήταν δυνατόν. Έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριμένες εκθέσεις από αυτού και έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένες δράσεις, κυρίως όσον αφορά τη προώθηση των συνεργειών, πολιτικοστρατιωτικών συνεργειών, καλύτερο συντονισμό των battle groups, την εκπαίδευση, και χρηματοδότηση, συνεργασία με βασικούς εταίρους και συγκεκριμένα το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, στηρίζουμε την ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε ήδη ε, από κοινού πετύχει πολλά. Η ύπατη εκπρόσωπος ε, για μία ακόμα φορά συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λισαβόνα την περασμένη, το περασμένο Σάββατο. Η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ αποτελεί σημαντικό ζήτημα όπως ε, χτες μόλις ε, ε, διατυπώθηκε στην διάσκεψη κορφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα και εφαρμόσουμε όλα τα πρακτικά μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν τη συγκεκριμένη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ και να εξασφαλίσουν όλους ιδιαιτέρως τη συνεργασία όταν και οι δύο είμαστε ανεπτυγμένοι στο ίδιο θέατρο. Ε, η Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος προσβλέπουν στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του σημαντικού αυτού θέματος πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, σε δεκάμιση. Κλείνουμε τώρα. Αύριο ξανά θα ξεκινήσουμε στις 9 με 1, 3 με 8.30 και 9 με 12 το βράδυ. Η ημερήσια διάδειξη είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ και έχει δημοσιευθεί κιόλας. Διακόπτεται η συνεδρίαση.